ζητήσει πρώτος να μιλήσω στη διαδικασία αυτή. Just a second, please. Και το έλεγξα... I'm Just sorry. a second, please. I want to finish. Και το έλεγξα... I'm sorry. You asked for a point of order. Yeah, I this is a point of floor. order and I would like to raise it and I would like to give me only 10... Ναι, είναι διαδικαστικό και 10 δευτερόλεπτα χρειάζομαι. Εντάξει, 10 δευτερόλεπτα χρόνος. Μετρήστε, 10 δευτερόλεπτα πρώτος... Well... Ten seconds, please. Είχα... Sir, the ten seconds are over. I'm sorry. Πέρασαν τα 10 δευτερόλεπτα, λυπούμε, λέει η Πρόεδρος. Micro. Micro.